Okay, wir legen mal los. So, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας καλησπερίσω στη σημερινή μας συνεδρίαση. Ε, ξέρω πως ε, αρκετοί συνάδελφοι έχουν προβλήματα με τους περιορισμούς λόγω του κορονοϊού και δεν ήταν δυνατόν να έρθουν σήμερα διότι είτε βρίσκονται σε καραντίνα είτε έμειναν στις πατρίδες τους. Όμως ε, και να έμειναν στο σπίτι τους ε, μπορούν επίσης να κάνουν το έργο του Κοινοβουλίου. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να έρθουν όλοι στις Βρυξέλλες, γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ. Καλησπέριζω επίσης και όσους μας βλέπουν μέσω της οθόνης τους. Από τον Απρίλιο έχει αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουμε και δεν βλέπω να αλλάζει σύντομα. Επομένως ε, υπάρχουν όντως κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές μας τις αίθουσε που έχουμε διαθέσιμες και τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να είναι δυνατό να μας παρακολουθούν όλοι από το διαδίκτυο, όμως ε, μια που δεν είμαστε τόσο πολύ άριθμοι σήμερα νομίζω ε, πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας ενημερώσω επίσης ότι στο Στρασβούργο θα παρέχεται διερμηνία από τις Βρυξέλλες έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ταξιδέψει πάρα πολλοί κόσμος στο Στρασβούργο. Το τμήμα πληροφορικής μας κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε βήμα-βήμα, αργά αλλά σταθερά να ε, λύσουμε όλα τα προβλήματα και τους ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να έχετε καλή διάθεση για να περάσουμε αμέσω στην ημερήσια διάταξη. Ε, θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω αν υπάρχουν σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Κάποιος από την αίθουσα ή από ε, το διαδίκτυο. Όχι. Ωραία λοιπόν. Εγκρίνονται λοιπόν ε, τα πρακτικά. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Από τις 3 μέχρι τις 4 παρατέταρτο θα γίνει κυκλισμένων των θυρών μία ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της ΕΤΕΠ σχετικά με τις ε, τρέχουσες εξελίξεις για την ε, επανεξέταση των διαδικασιών της ΕΤΕΠ για την καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω, όπως συνηθίζεται στις άλλες επιτροπές, όποιος επιθυμεί να παραστεί να είναι εγκαίρος. και να είναι στην ώρα του. Διαφορετικά θα πρέπει να μας αφήσει εγκαίρος. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Υπάρχουν αντιρρήσει ή κάποια σχόλια πάνω στα πρακτικά. Όχι. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, η απαλλαγή του 2018, Γενικός Προπολογισμός της Ένωσης για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα που εξετάζουμε εδώ είναι σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ο κορονοϊός έχει αναβάλει ε, τη διαδικασίες. Δεν ήταν δυνατόν να συναντηθούμε τους ε, περασμένους μήνες, όμως θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Στεχόφσκι για να μας ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις. Τόμας, μας ακούς? He seems to be Ο Τόμας φαίνεται πως έχει συνδεθεί, αλλά δεν είναι ακόμα εκεί. Γεια σας, γεια σας. Δύσκολο να σας δω πίσω από τις μάσκες. So we try to find... Ψάχνουμε λοιπόν τον εισηγητή μας. Θα σας εξηγήσω στο μεταξύ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να συναντηθούμε με το Συμβούλιο έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε μία ε, πιθανή συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής. Ελπίζουμε στα τέλη Οκτωβρίου η διαπραγματευτική ομάδα να καταφέρει να συναντηθεί και αν ε, καταφέρει να βρούμε τον εισηγητή θα σας τα έλεγε αυτός για να μην διαβάζω εγώ τις σημειώσεις του. Thomas is connecting. We work too quick for him. Ε, συνδέεται ο κύριος Σεντόφσκι. Φαίνεται ότι πάνε κάπως γρήγορα τα πράγματα για αυτόν. So Isabel, perhaps would you take the floor because you would be the... Θέλεις το λόγο Ιζαμπέλ, ε, διότι εσείς επόμενη ομιλήτρια και όταν συνηθεί ο Τόμας θα παρέμβει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορώ να παρέμβω τώρα, λέει η κυρία Γκαρθία Μουνιώθ και έτσι θα έχουμε, δώσουμε τον χρόνο στον κύριο Σερχόσκι να προετοιμαστεί. Λοιπόν, συμμερίζομαι με αυτά που είπατε στην αρχή της συνεδρίασης, ε, σας καλωσορίζω και εγώ όλους, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβλέπω όλους εσάς και εδώ από κοντά αλλά και τους υπόλοιπους μέσω της τεχνολογίας. Είναι δύσκολες, δύσκολες εποχές αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο ε, έκθεσης που παρουσιάζει ορθώς την κατάσταση σε ό,τι αφορά την απαλλαγή. Είναι πραγματικά απογοητευτικό ότι το Συμβούλιο δεν συνεργάζεται με την Επιτροπή μας, ε, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να μην εγκρίνουμε την απαλλαγή για άλλη μια φορά. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι αισιόδοξη και ελπίζω ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου, στην οποία ανήκω, και πραγματικά θέλω να χαίρομαι ιδιαίτερα που συμβαίνει αυτό, αποκοινούμε τον κύριο Συγητή και την πρόεδρο της Επιτροπής, της Επιτροπής μας, ε, Ελπίζω λοιπόν ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία για να μπει τέλος σε αυτή τη διαμάχη. Ελπίζουμε να γίνει αυτή η συνάντηση, εν Ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεση, αναφέρεται σε ορισμένα σημεία κλειδιά για την ομάδα μα, το υποχρεωτικό μητρό διαφάνεια, ο διαχωρισμό ε, των προπολογισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η νομοθετική διαδικασία και βεβαίω η ε, διαχείριση, η δημοσιονομική. Ε, δεν γίνεται αναφορά στο νέο οδηγό για ε, τους ιδιωτικούς σπόνσορες της Προεδρίας είχε ζητηθεί. Ε, το Συμβούλιο είχε απαντήσει θετικά. Ε, Αυτά δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ιζαμπέλ. Όλιβιέ, θα σου δώσω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω για το θέμα αυτό. Το γνωρίζει πολύ καλά. Από το 2009 ε, το θέμα το Κοινοβούλιο. Από τότε ε, δεν εγκρίνουμε την απαλλαγή, παρότι υπάρχει διαπραγματευτική ομάδα η δική μας με πολύ καλή θέληση ε, στη συζήτηση με το Συμβούλιο, δεν μπορούμε παρά να υπενθυμίσουμε αυτό που μας ε, που ανέφερε η Επιτροπή ΑΦΚΟ, ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν για να υπάρξει μια ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής, να, εφαρ, να εφαρμοστούν, να γίνουν σεβαστές όλες οι εφαρμοστές διατάξεις της συνθήκης. Εφόσον δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη, μιας και δεν έγινε και συνάντηση, δεν βλέπω πώς ε, μπορούμε να ε, εγκρίνουμε απαλλαγή σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ολιβιέ. Κύριε Κούς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι και εγώ που μπορούμε να συνεδριάσουμε επιτέλους, που ξαναβλεπόμαστε και μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Καλύτερα να μπορείς να βλέπεις ε, τον άλλο από το να κάνεις βιντεοδιάσκεψη. Σίγουρα είναι μεγάλη βελτίωση και έτσι κι αλλιώς ε, η βιντεοδιάσκεψη χάνει και υστερεί σε ποιότητα από το ζωντανό. Τώρα αυτή η ιστορία δεν έχει τέλος. Μπορεί να μην μας πιέζει ο χρόνος, όμως χρειάζεται να δουλέψουμε και να αναγνωρίσουμε ότι το κέντρο του προβλήματος, η ρίζα του προβλήματος είναι στην ουσία η περιφρόνηση που δείχνει προς τα εμάς ε, το Συμβούλιο, Περιφρόνηση προ το Κοινοβούλιο και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. Αυτό έχει συμβεί και στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και στα προγράμματα οικονομική ανάκαμψη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Ένα θεσμικό όργανο το οποίο είναι... Ε, ισχυρό, έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλά παρόλα αυτά ε, είναι σε αυτήν την θέση. Αγνοείται. Χρειάζεται οπωσδήποτε λοιπόν να βρεθεί μία λύση. Τώρα όσο για το αν θα βρεθεί έχω κάποιες επιφυλάξεις. Και σε τελική ανάλυση πρέπει να δούμε και τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, αν έχει οποιοδήποτε νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον ε, Μίκουλας προτού μιλήσει ο Τόμας. Ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο αρνείται να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο στη δικασία απαλλαγής εδώ και 10 χρόνια. Δεν έχει δείξει επικοδομητικό πνεύμα στη διαπραγμάτευση, οπότε δεν πρέπει και εμείς να χορηγήσουμε την απαλλαγή για το υπολογισμό του 2018. Ε, βεβαίως είναι ανησυχητικό ε, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ε, Πρωθυπουργού της Τσεχίας ε, και ταυτόχρονα είναι διευθυντής μιας επιχείρησης που χαίρει πολλών ε, χρηματοδοτήσεων, κοντιλίων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτά. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα φήμης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επιμείνω επίσης ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η, η προσβασιμότητα και η διαφάνεια σε επίπεδο Συμβουλίου ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής είπε ότι η έλλειψη διαφάνειας αποτελεί κακή διαχείριση. Το Κοινοβούλιο ζητεί εδώ και χρόνια τη δημιουργία ενός κοινού μητρώου διαφάνειας. Ήρθε η ώρα το Συμβούλιο να το αποδεχτεί επιτέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να βγάλετε τη μάσκα σας όταν μιλάτε έτσι ώστε να κάνετε και τη δουλειά των διερμηνέων πιο εύκολη διότι διαφορά, διαφορετικά δεν μπορούν να δουν ούτε καν ε, τα χείλη σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς με μάσκα, γι' αυτό λοιπόν επιτρέπετε να τη βγάλετε όταν παίρνετε το λόγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, Τόμας Δεχόφσκι. Νομίζω πως τώρα έχει συνδεθεί. Τόμας, μας ακούς? Jetzt. Ja, wir hören dich. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, καλησπερίζω λοιπόν από την Τσεχική Γερουσία και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Είναι καλύτερα να σας κάνω τα σχόλιά μου στα αγγλικά. Αξιότιμη πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εισηγητής για το ζήτημα αυτό και όπως ξαναβλέπω βεβαίως μετά το καλοκαίρι, ελπίζω να περάσετε ευχάριστα τις διακοπές σας όσο γίνεται πιο μακριά από το COVID. Θα είμαι σύντομος υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Ε, υπάρχει απαλλαγή του Συμβουλίου αλλά και της ΕΟΚΕ. Αναβάλαμε την έγκριση της απαλλαγής για το 2018. Υπάρχουν δύο σχέδια έκθεσης που περιλαμβάνουν ορισμένα ενδιαφέροντα νέα στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση που αναφέρεται στην έκθεση της απαλλαγής που ψηφίσαμε την Άνοιξη. Εν συντομία να επενθυμίσω το λόγο της αναβολής. Η απαλλαγή του Συμβουλίου αναβλήθηκε λόγω της υπάρχουσας κατάστασης. Το Συμβούλιο δεν συμμετέχει στην διαδικασία απαλλαγής εδώ και χρόνια και για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και για την ΕΟΚΕ λόγω του αποτελέσματος της έρευνας της Όλαφ Γιατί μη ηθική συμπεριφορά ενός μέλους της ΕΟΚΕ. Βεβαίως τώρα συζητάμε μόνο την απαλλαγή του Συμβουλίου και θα ξεκινήσω από αυτό. Η έκθεση για το Συμβούλιο επικεντρώνεται στα μελλοντικά βήματα που θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την υπάρχουσα κατάσταση και υπενθυμίζουμε και εν συντομία το τι συνέβη στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το εξή. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο, από, από, το, από την, συγγνώμη, από την διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου, να ξεκινήσει διαπραγμάτευση για τη διαδικασία απαλλαγή του Συμβουλίου, με το Συμβούλιο. Η διαπραγμάτευση από πλευράς Κοινοβουλίου γίνεται από την πρόεδρό μας, τη Μόνικα Χολμάιερ, ο πρώτος αντιπρόεδρος, η κυρία Ισαμπέλ Γκαρθία Μουνιώθ δηλαδή, και εγώ, ο οποίος είμαι συντονιστής και υπεύθυνο για την απαλλαγή για το 2018, για το σχετικό φάκελο. Έχει ενημερωθεί το Συμβούλιο σχετικά μέσω επιστολή και υπάρχει και ένα non-paper με τα κεντρικά σημεία. Πρέπει να γίνει σεβαστή η διαφορά μεταξύ των δύο διαδικασιών απαλλαγή. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να έχουν μια κοινή βάση στη συζήτησή τους για να μπορέσουν να οδηγήσουν, σε μια σύσταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο πρέπει να πάρθει μια απόφαση βεβαίως. Λόγω του κορονοϊού είναι δύσκολο να βρεθεί μια ημερομηνία για την πρώτη συνάντηση διαπραγμάτευσης. Μάλλον θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου αυτή η συνάντηση Και τώρα να δώσω ξανά το λόγο στις Βρυξέλλες. Ακούσω τη συζήτηση και μετά να κάνω κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη που άργησα. Κανένα πρόβλημα, μας Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι σκιώδες εισηγητές ήδη έχουν τοποθετηθεί υπάρχει σύπνη απόψεων. Τον Οκτώβριο θα προχωρήσουμε. Θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας κυρίως Βέλη στην ε, διαπραγμάτευση. Και ελπίζω να αποκτήσουμε επιτέλους μια ευκαιρία τουλάχιστον να ε, δώσουμε ένα αίσιο τέλος σε αυτή την ε, ιστορία. Μπορώ λοιπόν να περάσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον Τόμας για να σας ενημερώσει. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank. Θα μιλήσω αγγλικά για να καταλάβετε καλύτερα την προσέγγιση μου. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Ζιλ Γκυλάχ, το Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ΕΟΚΕ. Ο κύριος Αγγιλάρ αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ, τον κύριο Μπρουνέτη, που κολλείεται, δεν μπορεί να έρθει σήμερα, γιατί κάνει μια εγχείρηση. Του στέλνουμε λοιπόν θερμότατες ευχές ε, για γρήγορη ανάνυψη. Μετά τις ε, παρεμβάσεις και τις ενδεχόμενες απορίες ε, των Ευρωβουλευτών, ο κύριος Γκυλάρ θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Την Άνοιξη του 2020 έπρεπε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή, μας, στην Επιτροπή για το σχέδιο απαλλαγής για την ε, ΕΟΚΕ. το σχέδιο έκθεσης για την απαλλαγή για την ΕΟΚΕ. Και έπρεπε να εξετάσουμε και το γεγονός ότι η Όλαφ είχε υποβάλει μία έκθεση, καταλήγοντα στο συμπέρασμα ότι ένα ανώτερο στέλεχος της ΕΟΚΕ ήταν υπεύθυνο για κάποιες ενέργειες παρενόχλησης και σοβαρής ανάρμοστης συμπεριφοράς και παρά, Αποφασίσαμε λοιπόν να αναβάλουμε τη χορήγηση απαλλαγή στην ΕΟΚΕ προκειμένου να ζητήσουμε κάποιες πληροφορίες για τα μέτρα που ενδεχομένως έλαβε η ΕΟΚ για να διορθώσει ε, αυτά τα κακό κείμενα του συγκεκριμένου μέλους της. Στην, στο δεύτερο σχέδιο εκθεσής μου σας ενημερώνω για όλα αυτά τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Στις 16 Ιουνίου του 2020, η πρόεδρός μας, η κυρία Μόνικα Χολμάγερ και ο υποφαινόμενος λάβαμε επιστολή από το Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ με ένα κατάλογο των μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή μετά τις παρατηρήσεις στην απόφαση περί απαλλαγής. Η ΕΟΚΕ και ο πρόεδρος καταρχάς λαμβάνουν την έκθεση της ΟΛΑΦ και τις συστάσεις της ΟΛΑΦ στις 17 Ιανουαρίου του 2020. Η υπόθεση παραπέμπεται στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΟΚΕ, ε, αρμόδια για τη συμπεριφορά των μελών, στις 23 Ιανουαρίου του 2020. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει τα συμπεράσματά της στις 28 Απριλίου του 2020. Το λόγο μέλος ΟΚΕ καλείται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του ε, στις 12 Μαΐου του 2020 ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ καλεί το διευρυμένο Προεδρείο να υποβάλει σχόλια στις 27 Μαΐου του 2020. Ο ήχος του κυρίου Δεχόφσκη πραγματικά είναι πολύ προβληματικός, εν πάση περιπτώσει. Το Προεδρείο είχε μία κεκλεισμένα το θυρών τη διοίκηση παρουσία του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής με θέμα τη συμπεριφορά των μελών και παρουσία και των εκπροσώπων της Όλαφ που απάντησαν σε ερωτήσεις. Και στο τέλος, στο Προεδρείο της ΕΟΚΕ πήρε τι ακόλουθε αποφάσει με πλειοψηφία. Τα βασικά στοιχεία των αποφάσεων είναι ο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο μέρο ΕΟΚΕ ζητήθηκε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του πρόεδρου της ομάδας 1. Ε, ο συγκεκριμένος, ε, το συγκεκριμένο μέρο τη ΕΟΚΕ ε, ζητήθηκε να αποσύρει την αίτησή του για μια, και την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΟΚΕ. Επίσης, α, πελάγι όλων των δραστηριοτήτων που αφορούσαν διαχείριση ή ε, διοίκηση προσωπικού. Πέραν των αποφάσεων αυτών, η Ολάφ υπέβαλε, ολαφη υπεβαλε παρεπεμψε την υπόθεση μάλλον στις βελγικές, αρχές και τα εσωτερικά μέτρα της Επιτροπής, ε, της ΕΟΚΕ και τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής ανοχής κατά της παρενόχλησης. Επίσης, όλες αυτές οι σκέψεις και τα πορίσματα θα συμπεριληφθούν σε ένα διεξοδικό σχέδιο δράσης για το οποίο θα μας κρατάει ενήμερους η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Τώρα καλώ τους σκιώδεις ηγητές να μας παρουσιάσουν τις ε, παρατηρήσεις τους και κατόπιν να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΕΟ και τον κύριο Γκυλάρ. So, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ιζαμπέλ τώρα έχει τον λόγο σε σκιώδηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Γκυλάρ που ήρθε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής. Λυπάμαι που ο κύριος ε, Μπρουνέτη απουσιάζει. Ε, το ευχόμαστε σιδερένιο στο συντομότερο δυνατό. Ε, διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση μετά την υποβολή παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, για να καταλήξω συμπέρασμα αν θα πρέπει να εγκρίνουμε την απαλλαγή για το 2018. Έχω πολλές απορίες, φαντάζομαι θα προλάβετε να, να μου τις απαντήσετε όλες. Ε, ζητώ λοιπόν, ε, αν γίνεται, να τις υποβάλω γραπτός και να μου στείλετε τις απαντήσεις το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω να είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Τι γίνεται με τον κύριο Κράτσεκ σε ό,τι αφορά την προεδρία της ομάδας 1 και την υποψηφιότητά του ε, για την Προεδρία της ΕΟΚΕ. τι μέτρα έχουν ληφθεί για να αποφευθεί οποιαδήποτε επαφή του κ. Κράτσικ με τη γραμματεία και το προσωπικό του, της ομάδας 1 όπως πρότεινε τον Ιούνιο του 2020 η ΟΛΑΦ έγιναν ε, κάποιες ενέργειες ώστε να αντικατασταθεί ο κύριος Κράτσικ από την Προεδρία της Ομάδας 1 και να αποσυρθεί η υποψηφιότητά του από, για την Προεδρία της ΕΟΚΕ. Σε περίπτωση που δεν δεχτείτε τα απορίσματα του Προεδρείου και δεν επιλέξει το Προεδρείο άλλον υποψήφιο για την Προεδρία της ΕΟΚΕ, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η ΕΟΚΕ για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ε, σε ό,τι αφορά τις της ΟΛΑΦ, η ΕΟΚΕ μας ενημέρωσε ότι έλαβε κάποια συμπληρωματικά μέτρα για να προσφέρει διοικητική ε, και ψυχολογική αρρωγή στα μέλη της γραμματείας της ομάδας 1. Ποια ήταν αυτά τα μέτρα. Εφαρμόστηκαν και στους καταγγέλλοντες και στα θύματα. Τον Ιούλιο του 2018, ο Διευθυντής ε, Ανθρωπίνων Πόρων έλαβε πολλές καταγγελίες για παρενόχληση του κ. Κάτσικ ε, και μάλιστα έγινε και μια αναφορά προς τη ιατρική υπηρεσία από τη γραμματεία της ομάδας 1. Και μάλιστα έχει, ε, και τον Ιούνιο μια έκθεση προς τον ΟΛΑΦ. Ε, έχουμε μείνει πίσω στο χρόνο, έχουμε μεγάλη πίεση, γι' αυτό και οι σκιώδεις ηγητές έχουν μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή τους. Παρακαλώ, χρόνου φίδου. Ναι, είμαι συνοπτική. Το θέμα είναι ότι έχω πολλές ερωτήσεις προς τον πρόεδρο της ΕΟΚΕ. Γι' αυτό ζήτησα να τη στείλω γραπτός τις περισσότερες. Περιορίστηκα σε ορισμένες μόνο. Έπρεπε να στείλετε αυτή την πληροφορία στην ΟΛΑΦ με βάση τον εσωτερικό, το καταστατικό του προσωπικού και τη διοργανική συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, μόνο τον Νοέμβριο του 2019, ένα χρόνο μετά, πέρασε και, περίμενε η ΕΟΚΕ για να υποβάλει αυτή την έκθεση και στην ΟΛΑΦ. Ε, η νομική υπηρεσία έκανε κάποια γραμμάτευση πέρα του κυρίου Κράτσεκ και σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Προβλέπονται συγκεκριμένες αλλαγές στην ε, διαδικασία την πειθαρχική, μια και οι ισχύουσε διατάξεις φάνηκαν ανεπαρκείς για την περίπτωση την υπόθεση του κυρίου Κράτσικ. Επίση, η γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία έχει νόημα όταν έχει κάποια προστιθέμενη αξία. Με ποια κριτήρια όμω κρίνεται αν είναι σκόπιμη η διαβούλευση με την νομική υπηρεσία. Επίση, πώ θα εξασφαλίζεται η γνωμάτευση νομική υπηρεσία για αποφάσει που ε, αφορούν την μη χορήγηση της απαλλαγής. Εδώ και χρόνια έχουμε ε, ζητήσει διοντολογικό κώδικα ε, των μελών της ΕΟΚΕ. Χρειάστηκε να γίνουν αυτές οι καταγγελίες της παρενόχλησης για να εφαρμοστεί επιτέλους αυτός ο διοντολογικός κώδικας. Γιατί καθυστερήσατε τόσο. Με αγροκοιτάζει η Πρόεδρος, γι' αυτό και τις... Ναι, σας παρακαλώ ε, πραγματικά να τα κάνετε αυτά πριν την ε, συνεδρίαση, διότι δεν μπορούμε να αφιερώσουμε μισή ώρα για ερωτήσεις πριν τη συνεδρίαση και να υπάρχει μισή ώρα για απαντήσεις. Αν θέλουν να μιλήσουν όλα τα μέλη, δεν θα προλάβουμε. Ας το κάνουμε όπως έχουμε συνηθίσει, δηλαδή να στείλουμε γέρος ερωτήσεις στην ε, ΕΟΚΕ και επίσης τα μέλη των ε, επιτροπών δεν είναι υπάλληλοι και δεν ε, υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Αυτά είναι θέματα δικαστηρίου και εάν θα δικαιωθεί ο κατηγορούμενος ή όχι. Οι πειθαρχικές διαδικασίες αφορούν μόνο τους υπαλλήλους υπαλλήλους της ΕΟΚΕ. Από όσο γνωρίζω, ε, λοιπόν, ε, θα ήθελα να προτείνω να ζητήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα, στον φάκελο της Όλαφ, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα συνεδριάσουμε να εστιάσουμε στα ουσιώδη. Εάν καταφέρουμε να δούμε τις ε, αναφορές και τα αρχεία, τότε θα καταφέρουμε να σχηματίσουμε και καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη άποψη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απευθύνετε την ερώτησή σας κατευθείαν στην ε, ΕΟΚΕ και να συνεχίσουμε με την συνεδρίαση γιατί μας πιέζει αρκετά ο χρόνος. Και εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Χάν, ο οποίος ήδη περιμένει για το επόμενο θέμα. Ολιβιέ, ο λόγος ξανά σε σένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και εγώ θέλω βεβαίως να χαιρετήσω την συνειδητοποίηση ε, της, του, του, ε, της ΕΟΚΕ, της όλης κατάστασης και της προσπάθειας που έχει κάνει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει κάποια, κάθε μορφή ε, παρενόχλησης. Όμως ε, η έκθεση της Όλαφ είναι πραγματικά καταιγιστική ε, για αυτές τις ε, υποθέσεις ε, παρενόχλησης και πλέον έχει αναλάβει και βελική δικαιοσύνη. Βεβαίως ε, υπάρχει πάντα η, ε, η αρχή ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι αποδείξει στον αντίου, όμως ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το παρόν και το μέλλον του ε, κατηγορούμενου. Όμως ένα άρθρο στον τύπο αναφέρεται στο θέμα αυτό με ανησυχητικό τρόπο. Το Προεδρείο της ΕΟΚΕ, από ό,τι φαίνεται, πήρε μια σειρά από αποφάσεις στις 9 Ιουνίου και από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει ο τύπος χθες, το, το εν λόγω άτομο, από ό,τι φαίνεται, αποφάσισε 28 Αυγούστου να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του. Παρότι, παρόλα αυτά που, είχε, που, του είχε, που του είχαν υποθεί από το Προεδρείο της ΕΟΚΕ. Οπότε και εγώ αναρωτιέμαι, όπω οι συνάδελφοι, πριν λοιπόν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση σε ό,τι αφορά την απαλλαγή για το 2018, θα πρέπει να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα για τι αποφάσει που έχουν πάρθει, διότι από ό,τι φαίνεται αυτέ οι αποφάσει δεν έχουν εφαρμοστεί. Υπάρχει το θέμα της αντίδρασης του ενδιαφερομένου, ο τρόπος με τον οποίο, ε, από ό,τι φαίνεται, είναι ο μόνος υποψήφιος για την Προεδρία της ΕΟΚΕ, τι γίνεται με τη διαδικασία αυτή, μπορεί να ξανανοίξει. Ε, μια σειρά λοιπόν από ερωτήματα που πέρα από τα μέτρα που έχει πάρει η ίδια η ΟΚΕ, θέτουν το ζήτημα του κατά πόσο οι αποφάσεις αυτές που πάρθηκαν έχουν εφαρμοστεί. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ ευχαρίστω να με πείσουν, να με πείσει κάποιο το αντίθετο. Ε, να μας εξηγήσει η ΕΟΚΕ ποια είναι ακριβώς η κατάσταση αυτή τη στιγμή διότι αυτό το άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες, ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα χάος που υπάρχει στην ΕΟΚΙ αυτή τη στιγμή. Χάος. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε σήμερα εμείς να πάρουμε θέση για την απαλλαγή για το 2018. Ευχαριστούμε πολύ, Ολιβιέ. Έχετε θέσει όλοι πολύ σωστές ερωτήσεις και το θέμα αυτό είναι δύσκολο για μας. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε, ε, διότι παρότι δεν είμαστε αρμόδιοι για τα θέματα παρενόχλησης, είμαστε αρμόδιοι για θέματα προϋπολογισμού και απαλλαγής. Και έχω αμφιβολίες, οφείλω να ομολογήσω, για το ε, τι θα γίνει και αν θα καταφέρουν να απαντήσουν τις ερωτήσεις μας. Γιώχιμ Κούς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που είναι σαφές από την όλη διαδικασία είναι ότι τίποτα δεν είναι σαφές. Διαφο... Και γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Και θα πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει έτσι ώστε αργότερα το φθινόπωρο να μπορέσουμε να ε, συνεχίσουμε την ε, δουλειά μας, να απαντήσουμε αυτά τα αναπάντα ε, ερωτήματα. Χρειάζεται όμως σαφήνεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει όμως να αποφασίσουμε σύντομα, λέει η κυρία Χολμάιερ, όπως γνωρίζετε μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να έχουμε κάποια απάντηση να δώσουμε θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν, για παράδειγμα, εξαιτία ε, ελλείψεων δεν μπορούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή, διότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι λίγος. Η προθεσμία μας λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου και πρέπει μέχρι τότε να έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε. Ή θα χορηγήσουμε την απαλλαγή, όμως ε, θα πούμε ότι θα παραμείνει ανοιχτό το θέμα στην επόμενη απαλλαγή ή δεν θα χορηγήσουμε απαλλαγή. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν με τον εισηγητή τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Ε, δυστυχώς ε, δεν έχουμε χρονικό περιθώριο για να περιμένουμε εξηγήσει. Όμως το ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε είναι σαφές. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Νίκολας Πέτς. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα στην αρχή να συγχαρώ ε, την ε, ταχύτητα με την οποία η ΕΟΚΕ αντιμετώπισε το θέμα. Ο κύριος Κράφτσικ παρετήθηκε από πρόεδρος της ομάδας 1 και το σίγουρο είναι ότι δεν, ε, δεν επιτρέπεται να κριθεί ένοχος από την Όλαφ πρόεδρος ομάδας της ΕΟΚΕ. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων και του γεγονότος ότι ο κύριος Κράφτσικ καρνείται να παρετηθεί και δεδομένου ότι δίωκεται από τις βελγικές αρχές, εγώ δεν μπορώ να χορηγήσω απαλλαγή στην ΕΟΚΕ. Ε, η απόφαση που λήφθη από το Προεδρείο έχει ως αποτέλεσμα ο κύριος Κράφτσικ να συνεχίσει να είναι υποψήφιος ε, για την ε, επόμενη Προεδρία της ΕΟΚΕ, ενώ βρίσκεται υπό διερεύνηση από, από τις αρχές. Γι' αυτό λοιπόν η απόψη μου είναι αυτή που σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Η έχει ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκυγιάρ, Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων και ε, Δημοσιονομικών Θεμάτων. Σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι και να απαντήσετε γραπτά στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Μέχρι τις 10 ε, Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Σίγουρα θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα μέχρι τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να λάβουμε μια εμπεριστατωμένη ε, απόφαση. Όμως ε, θα σας δώσω τώρα αμέσως το λόγο για να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, αλλά και τα μέλη που πήραν το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Βεβαίως ε, ευχαριστώ να απαντήσουμε και γραπτός ε, στα ερωτήματα που θα λάβουμε. Θα επικεντρωθώ στα κεντρικά σημεία εδώ, να δώσω κάποιες απαντήσεις ε, σε σχέση με αυτά που άκουσα σήμερα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η αναφορά σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε χθες. Θέλω να σας ενθαρρύνω να διαβάσετε τη δήλωση του Προεδρείου της ΕΟΚΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ίδιο μέσο επικοινωνίας, το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Εκεί θα βρείτε μια σειρά από απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Τι έχουμε κάνει λοιπόν μετά την έκθεση της Όλαφ. Έχουμε αναλάβει μια σειρά από ενέργειες, από δράσεις απόλυτη συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΟΚΕ βέβαια, βοήθεια και προστασία των θυμάτων, πλήρης εφαρμογή της σύστασης της Όλαφ για να μην υπάρξει ε, νέο, νέο, νέο τέτοιο κρούσμα στο μέλλον, απόλυτη συνεργασία με τις ε, δικαστικές αρχές του Βελγίου για την υπόθεση αυτή, ενημέρωση κατά διαφανή τρόπο των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης ε, και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, τον Μεσολαβητή, την Όλαφ ε, με βάση βεβαίως τα καθήκοντά μας, την υποχρέωσή μας στην πλαίσια διαθυμικής συνεργασίας και βέβαια πρέπει να, να αντλήσουμε και κάποια διδάγματα, να γίνει μια αξιολόγηση σε βάθος του υπάρχοντος πλαισίου κατά της ε, παρενόχλησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Ό,τι αφορά την αποφάση του Προεδρείου που πάρθηκε στις 9 Ιουνίου και που ανέφεραν διάφοροι ομιλητές, θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση εφαρμόστηκε πλήρως από την ε, ΕΟΚΕ. Δεν υπάρχει κανένα χάος στην ΕΟΚΕ. Αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω εγώ. Και ως επικεφαλής των ανθρωπίνων πόρων στον ΕΟΚΕ, πρέπει να σας πω ότι ο ενδιαφερόμενος ε, πλέον δεν έχει πλέον κανένα καθήκον στην πλαίσια της διαχείρισης, ε, της διοίκησης. Όλα αυτά τα έχουν αναλάβει είτε ο Γενικός Γραμματέας, είτε εγώ. Ε, είναι σαφείς οι οδηγίες που έχουν δοθεί προς, το, προς την κατεύθυνση αυτή. Σας καλώ για άλλη μια φορά να διαβάσετε τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ, την οποία μπορώ και να σας ε, στείλω και μπορείτε να βρείτε όμως ήδη στον τύπο σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η σύντοση της ΕΟΚΕ στην Ολομέλεια στις 28 Ιουνίου αποφάσισε να άρει την ασυλία του, του μέλους αυτού και να προσφέρει ε, νομική ενίσχυση σε, ε, στο, πρώην, στο πρώην μάλιστα της ΕΟΚΕ, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, ε, για τα θύματα αυτών των ενεργειών. Σε ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση, να θυμίσω ότι όπως γνωρίζετε τα μέλη της ΕΟΚΕ ορίζονται από τα κράτη-μέλη και επισήμως ε, τοποθετούνται από το Συμβούλιο. Εκεί η ΕΟΚΕ δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τελικά η ολομέλεια της ΕΟΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο για την εκλογή του Προέδρου. Τέλος, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέλος, εξακολουθεί να είναι μέλος της ΕΟΚΕ και του Προεδρίου. Όπως εξήγησα, αυτό είναι κάτι ε, το οποίο εμείς δεν ελέγχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κάτι άλλο που αναφέρεται στη δήλωση του Προέδρου, ε, υπάρχει άλλο ένα μέλος της ΕΟΚΕ που είναι υποψήφιο για την Προεδρία οπότε υπάρχει τουλάχιστον ακόμα ένα όνομα και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις από αυτού. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω μάλλον στα όλα τα ερωτήματα τα οποία ανέφεραν οι σκιώδεις ε, Ευχαρίστως ε, να απαντήσω γραπτός βεβαίως. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι η ΕΟΚΕ πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει την υπόθεση αυτή και αποδείξαμε και το πόσο δεσμευόμαστε σε αυτή την πολιτική μηδενικής ανοχής όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, που συμμετείχατε στην ε, σημερινή συζήτηση. Σίγουρα θα σας ε, στείλουμε τις ερωτήσεις γραπτά. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω και τον ε, Τόμας Δεχόσκι. Είστε ακόμα στην γραμμή ή θέλετε να πείτε κάποια λόγια για το τέλος. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούμε κύριε Στεχόφσκι. Δεν υπάρχει ήχος. Η σύνδεση είναι πολύ κακή ούτως ή άλλως από την αρχή. Με ακούτε τώρα. Σας, ακού, σας ακούμε τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ήταν συναρπαστική συζήτηση. Είμαι πολύ περήφανος γιατί ε, ήταν πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις και οι απορίες των σχεδόν εισηγητών και τους ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό και την έντονη τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση με την ΕΟΚΕ και ε, άλλα θέματα που είναι σημαντικά για τη χορήγηση της απαλλαγής. Ο κύριος Γκελάρ είχε δίκιο σε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε την ΕΟΚΕ, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η στάση που κρατήσατε και η απόλυτη διαφάνεια που δείξατε στην απάντηση των ερωτήσεων. Θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η σημαντική συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες λίγη τη Δευτέρα στις 10 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ η ψηφοφορία και για τα δύο θέματα θα γίνει την 1η Οκτωβρίου του 2020. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να παραμείνετε ασφαλείς όχι και βλαβή Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε στείλει τις ερωτήσεις σε εμάς μέχρι αύριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τις προωθήσουμε στην ΕΟΚΕΒ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ε, να πω πως χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ τον Επίτροπο Γιωχάννης Χάν και τον Γενικό Διευθυντή Ήταλα. Πού είστε, να εδώ είστε. Καλώς ήρθατε. Κρύβεστε όλοι, σας κρύβουν και οι μάσκες, δυσκολεύομαι να σας δω. Να καλωσορίσω και τον Γιάνν Μούλτερ, ο οποίος έχει συνδεθεί μαζί μας Σας ευχαριστώ πολύ. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Μούλτερ είχα και ένα τύχημα. Όχι ότι έχει καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων. Να σας πω λοιπόν ε, πολύ σύντομα ότι το θέμα αυτό αφορά την αναδιάρθρωση της Όλαφ. Για εμάς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού η Όλαφ είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία. Εδώ Πάλι έχουμε συναντήσει προβλήματα με το Συμβούλιο. Η Όλαφ δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία και ορισμένους ε, τραπεζικούς ε, λογαριασμούς για να ασκήσει το έργο της. Ε, να, να σας διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, διότι είναι έργο μας και έργο σας να ελέγχουμε τα πράγματα όταν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια παρατυπία. Το έργο σας είναι να ακολουθείτε την πορεία του χρήματος και πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Όταν λοιπόν σας κόβουν και σας εμποδίζουν, αυτό καταλαβαίνω πόσο ενοχλητικό είναι. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω λοιπόν άλλη μία φορά. Σας ευχαριστώ που ε, είστε εδώ. Έχετε ασχοληθεί ενεργά με το ε, θέμα. Η αναδιάρθρωση της Όλαφ έχει άμεση σχέση και με τη νέα σχέση της με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξουν ε, σύνδεσμοι μεταξύ των δύο υπηρεσιών Δυστυχώς και ε, θα σας δώσω τον λόγο αφού πρώτα σας παρακαλέσω να δώσετε τη στήριξή σας στον Όλαφ έτσι ώστε να μην ε, χρειαστεί να γίνουν περικοπές, οι περικοπές που έχουν προταθεί. Και να σας ενημερώσω επίσης στα αγγλικά ότι μαζί μας είναι και ένας εκπρόσωπος της ε, Κεντρικής Επιτροπής Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Κριστιανό Σεμπαστιάνη, ο οποίος ε, θα έχει το τη δυνατότητα να σχολιάσει εφόσον το επιθυμεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα προσωπικού. Επίσης, ο Ματίας Βίλ, εκπρόσωπος ε, του οργανισμού ε, της ε, Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης είναι μαζί μα, ε, ο οποίο είναι επίση στη θέση να απαντήσει σε ερωτήσει σας. Θα δώσω τώρα το λόγο ευθύ αμέσω στον Επίτροπο Χάν. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσπίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να εξασφαλίσουμε ένα, μια ισχυρή Όλαφ, μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, κάτι που σημαίνει και την απαραίτητη στελέχωση και ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει τις ε, διαπραγματεύσεις για το ΠΔΛΤΑΠ. Θα δούμε ποια είναι η τελική έκβαση των συζητήσεων. Πάντω σα ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση να λάβω μέρο σήμερα στη συζήτηση για, μετά την πρόσφατη αναδιοργάνωση της ε, υπηρεσία καταπολέμη απάτη στι 16 Ιουνίου του 2020. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν και η πρόσφατη πανδημία θα έλεγα είναι καλό παράδειγμα, όχι καλό με την έννοια ότι ήταν ε, χρήσιμο, αλλά πραγματικά ενδεικτικό πόσο μπορούν να αλλάξουν ραγδαία οι προκλήσει. Και πολύ φοβάμαι ότι η συγκεκριμένη πρόκληση τη πανδημία δεν πρόκειται να εξαφανιστεί πολύ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να προσαρμόζεται γοργά, ακόμη και στην εσωτερική τη διοργάνωση. Οι πόροι μας θα πρέπει να παραμείνουν στρατηγικά ευθυγραμμισμένοι προ τι πολιτικέ και επιχειρησιακέ μας προτεραιότητε και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και σε αυτό το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τη διακριτική της ευχέρεια για να αναδιοργανώσει τι γενικέ διευθύνσει τη, όποτε είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, και ακολουθώντας τις καθευθυντήριες γραμμές ε, για τα οργανογράμματά της. Η αναδιοργάνωση της ΟΛΑΦ ήταν το αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής εκτενέστατης διαδικασίας ε, και εντός της ΟΛΑΦ αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι προετοιμασίες αυτές ε, κράτησαν ένα ολόκληρο χρόνο και με βάση τις πάγιες διαδικασίες το εγχείρημα αυτό διεξήχθη σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων διαχειρίζεται τη διαδικασία λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση των οργανωτικών δομών σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία και άλλες ε, ενδιαφερόμενες και αρμόδιες ομάδες. Το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε τη νέα οργανωτική δομή της ΟΛΑΒ στις 20 Μαΐου και τέθηκε σε ισχύ από τα μέσα Ιουνίου. Αυτό είναι ένα πάγιο και δρεωμένο δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως και οποιασδήποτε άλλη διοίκηση Και δεν είναι μυστικό κάτι τέτοιο. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνεχίζει ε, να υπόκειται στην εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτική βάση για τις δραστηριότητές της. Στην ε, ειδική περίπτωση της ΟΛΑΒ, το Κοινοβούλιο συμμετέχει ως παρατηρητή στη Συμβουλευτική Επιτροπή ε, των Διορισμών για την επιλογή της νεπαγούς θέσης του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΟΛΑΒ, που ήδη συμπεριλαμβάνεται στο νέο οργανόγραμμα της ΟΛΑΒ. Ο σκοπό τη νέα αναδιοργάνωση τη ΟΛΑΒ είναι να βελτιστοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν ε, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα και τη υπηρεσία ε, ω Γενική Διεύθυνση αλλά και των ε, ανεξάρτητων ερευνητικών τη δραστηριοτήτων. Όπω ξέρετε, είναι περιορισμένη η πόρη τη ΟΛΑΦ, οπότε θα πρέπει να αξιοποιούνται στο έπακρο. Κάτι τέτοιο είναι η προπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε αλλαγή στην οργάνωση και τη δομή τη. Ε, η αναδιοργάνωση αυτή έχει στόχο να ετοιμάσει την ΟΛΑΦ να ξεπεράσει τι νέε προκλήσει στην καταπολέμηση τη Απάτη, να προσαρμοστεί στις νέε πολιτικέ προτεραιότητε τη Επιτροπή Φοντερ Λάιν, να εφαρμόσει τη στρατηγική καταπολέμηση απάτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνεργαστεί αποτελεσματικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε λίγο, ο Γενικό Διευθυντής της ΟΛΑΦ, ο Βίλε Ήταλα, θα σα ε, παράσχει πιο διεξοδικέ πληροφορίε για την αναδιοργάνωση τη ΟΛΑΦ θα σας παρουσιάσει τις αλλαγές στην δομή της υπηρεσίας αυτής και θα σας εξηγήσει το πώς οι αλλαγές αυτές θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Και μάλιστα ήταν πολύ επίκαιρη αυτή η ανοδιοργάνωση, γιατί ετοιμαζόμαστε να επενδύσουμε πρωτοφανή ποσά στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να βαθμίσουμε τη συλλογική μας δράση για να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Είμαι πεπισμένο ότι η νέα δομή τη ΟΛΑΦ είναι πλήρω εξοπλισμένη για να ανταπεξέλθει στην εντολή τη και να προστατεύσει τον κοινοτικό προπολογισμό ακόμη πιο αποτελεσματικά και στο σκέλο των ερευνητικών δραστηριοτήτων και σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε τη πολιτική. Σα ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Ιταλό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τη νέα οργανωτική δομή της ΟΛΑΦ που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουνίου του 2020. Ε, θα σας μιλήσω σήμερα για το πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ΟΛΑΦ να σταθώ σε μερικές βασικές αλλαγές της δομής μας και να σας εξηγήσω επίσης γιατί αυτές οι αλλαγές θα εξασφαλίσουν μια ενίσχυση της ΟΛΑΒ στο μέλλον. Γιατί λοιπόν έγινε αυτή η αναδιοργάνωση πρώτα απ' όλα. Όπως γνωρίζετε όλοι, η ΟΛΑΒ ερευνά απάτες κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού και στο σκέλος των δαπανών και στο σκέλος των εσόδων. Επίσης, διερευνά και καταγγελίες ε, σοβαρών παραπτωμάτων και ανάρμα συμπεριφορά ε, του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των κοινωτικών θεσμικών οργάνων. Και μάλιστα η εντολή αυτή έμεινε απαράλλαχτη από τότε που ιδρύθηκε η υπηρεσία το 1999. Από την άλλη πλευρά, το έργο, το έργο μας κατά την εφαρμογή αυτής της εντολής και την εκτέλεσή της ε, αναπτύ, ανα, εξελίσσεται διαρκώς. Οι απαταιώνε δυστυχώς ε, μαθαίνουν πολύ γρήγορα και είναι πολύ πιο ευρηματικοί από ό,τι φανταζόμαστε. Η αποτελεσματική προστασία του κοινοτικού προπολογισμού σημαίνει επενδύσεις σε συνεχή προσαρμογή των εμπειρογνώσεων μας και των ε, εργαλείων μας στα νέε τάσεις και όλο πιο περίπλοκα συστήματα απατών. Και μάλιστα σε όλα αυτά τα χρόνια επενδύσαμε τα συλλογικά μας κονδύλια σε διάφορους τομείς ανάλογα με τις ε, νέες πραγματικότητες και σε ευθυγράμμιση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια υπηρεσία που ε, ερευνά και παρακολουθεί το χρήμα, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πρέπει και ο τρόπος που εστιάζουμε να τροποποιείται αντίστοιχα με τις ανάγκες. Όπως και οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, ε, μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας και αφιερώνουμε χρόνο στο να εντοπίσουμε τους τομείς που επιδέχονται βελτιώσει στο έργο μας. έτσι έχουμε τακτικά αναδιοργανώσεις της ΟΛΑΦ, όπως και άλλων υπηρεσιών της Ένωσης. Μάλιστα, έγιναν 20, 8 ε, συγγνώμη, τέτοιες αναδιοργανώσεις τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας της ΟΛΑΦ. Και όλες αυτές οι αναδιοργανώσεις είχαν τους δικούς τους σκοπούς και αντανακλούσαν το συγκεκριμένο πλαίσιο των, της λειτουργίας της ΟΛΑΦ. Και τον Ιούνιο έγινε η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας ε, με τρία βασικά μελήματα. Καταρχήν να καταστήσουμε την Όλαφ ε, ε, κατάλληλη για το μέλλον, κάτι που σημαίνει πρώτα απ' όλα εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα αναλάβει τη λειτουργία της από φέτος. Και μάλιστα για μια διεξοδική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στενή συνεργασία της ΟΛΑΦ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, έχει ύψη στη σημασία. Δεύτερο μέλημα, να προσαρμόσουμε το έργο της υπηρεσίας μας στις νέες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Φοντερ Λάιαν. Επικεντρωνόμαστε στην καταπολέμηση ε, και της περιβαλλοντικής δαπάνης, ε, απάτης και της απάτης στα τρόφιμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την, τελ, την Τελωνιακή Ένωση και να συμβάλλουμε στον μηχανισμό του κράτους δικαίου ε, σε σχέση και με το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτο μέλημά μας είναι να προετοιμάσουμε την Όλαφ να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και τάσεις στην καταπολέμηση των καθώς και νέα είδη απάτης που μπορεί να δημιουργηθούν στα πλαίσια των νέων ε, χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων και να εφαρμόζουμε φυσικά και τη νέα στρατηγική κατά τη απάτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα τη υπηρεσία μα και ω ανεξάρτητη ερευνητική υπηρεσία που εντοπίζει απάτε, αλλά και ω υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για την πρόληψη των απατών. Επίσης, η αναδιοργάνωση αυτή προετοιμάζει το έδαφος για να γίνουμε μια πιο ευέλικτη και σβέλτη οργάνωση. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Γενικός Διευθυντής της ΟΛΑΦ τον Αύγουστο του 2018, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από την προσήλωση του προσωπικού και τα αποτελέσματα που έχουμε υλοποιήσει. Ταυτόχρονα διαπίστωσα ότι κάποιες πτυχές του έργου μας μας εμπόδιζε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό της ΟΛΑΦ. Από την αρχή, ένα, μια θεμελιώδης πτυχή της διαδικασίας αναδιοργάνωσης ήταν η διαβούλευσή μου με τους υπαλλήλους της ΟΛΑΦ, με το προσωπικό της ΟΛΑΦ. Και μάλιστα το σεμινάριο προσωπικού που οργανώσαμε το Μάιο του 2019 μας επέτρεψε να συζητήσουμε τα βασικά εμπόδια, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες του προσωπικού και το πώς ε, η ΟΛΑΦ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική υπηρεσία. Και σε άλλες εσωτερικέ συζητήσεις που ακολούθησαν στην ΟΛΑΦ, συναντήθηκα με όλα τα μέλη του προσωπικού, είτε στις μονάδες τους, είτε και σε άλλη ευκαιρία. Πάντως, ε, θέλαμε μια νέα ΟΛΑΦ που θα είναι κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ε, και στις προσδοκίες των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ίδιου του προσωπικού της ΟΛΑΦ. Και ήδη διαπιστώνω ότι τα καταφέραμε και το έχουμε επιτύχει. Το βασικό συμπέρασμα από τις συζητήσεις που είχαμε του υπαλλήλους της ΟΛΑΦ ήταν η ανάγκη να βελτιώσουμε την ε, συνοχή και, την, ε, και το συντονισμό μεταξύ μονάδων που ενεργοποιούνται σε παρόμοιους τομείς. Τώρα βλέπετε το νέο οργανόγραμμα της ΟΛΑΦ και θα ήθελα να, να σας ξεναγήσω στις ε, βασικές αλλαγές που εφαρμόσαμε προκειμένου να βελτιώσουμε το έργο μας. Όπως βλέπετε από το νέο οργανόγραμμά μας, οι μονάδες πολιτικής ε, της ΟΛΑΦ ε, συνδέονται καλύτερα με τις ερευνητικές μονάδες της ΟΛΑΦ. Αυτό ήδη είχε θετικό αντίκτυπο, γιατί ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των διαφορών μονάδων και τις ανταλλαγές μεταξύ των μονάδων προκειμένου να έχουμε πιο εκτενή εντοπισμό απάτης και πρόληψη της απάτης. Επίσης, ε, ε, αξιοποιούμε καλύτερα αυτό το υβριδικό καθεστώς που έχουμε, που καλύπτει και έρευνες και πολιτική καταπολέμησης ε, απάτης, ενώ εξασφαλίζει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των, της διπλής αυτής λειτουργίας της ΟΛΑΦ. Οι νέες, για δαπάνες, ε, έσοδα και διεθνείς επιχειρήσεις, το Κέντρο Γνώσης κατά της ε, απάτης και γενικών υποθέσεων, μαζί με την ε, δημιουργία μιας θέσης αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, θα εξασφαλίσουν ότι οι τάσεις που εντοπίζονται από τις ερευνητικές ομάδες θα εντάσσονται στο έργο των μονάδων πολιτικής και των νομοθετικών μονάδων. Θα εξασφαλίσει συνέργειες και θα εξορθολογήσει το έργο μας προκειμένου να υλοποιήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των εργασιών μας. Ο τομέας επικοινωνίας επίσης ε, συγκεντρώθηκε και τέθηκε στη δική υπό τη δική μου ευθύνη, εξασφαλίζοντας καλύτερη σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς και πιο συνεπή ε, και συνεκτική επικοινωνία με τους πολίτες, τον τύπο και άλλα θεσμικά όργανα και φορείς. Επίσης, συστήσαμε μια ειδική ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση, προκειμένου να εξορθολογήσουμε, να συγκεντρώσουμε και να παρακολουθήσουμε τη συνέχιση που θα δοθεί στις συστάσεις που θα εκδώσουμε. Έχουμε ε, λάβει υπόψη την ανάγκη να ενισχύσουμε την παρακολούθηση των δικαστικών συστάσεων από την ΟΛΑΦ Κάτι που επισήμανε επανειλημμένω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ομάδα αυτή εργασία για την παρακολούθηση θα συγκεντρώνει πληροφορίε για την εφαρμογή όλων των συστάσεων τη ΟΛΑΒ και θα αναλύει τα αποτελέσματα προκειμένου να δει αν οι προσπάθειές μας αποφέρουν καρπού. Η αναδιοργάνωση λοιπόν που έγινε δεν ήθελε μόνο να βελτιώσει τις εργασίες μας. Η νέα δομή της ΟΛΑΦ έχει στόχο να προετοιμάσει την υπηρεσία μας για τις νέες προτεραιότητες και το νέο τοπίο καταπολέμησης της απάτης που χαρακτηρίζεται από την ίδρυση και της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης που υιοθετήθηκε πέρυσι. Και μάλιστα ε, βλέπουμε ότι η νέα οργάνωση πραγματικά λαμβάνει υπόψη αυτές τις ανάγκες. Όλα τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπίπτουν πια σε μία ενιαία μονάδα. Η Όλαφ θα συνεχίσει να ερευνά στις χώρες αυτές όπως το κάνει και σήμερα, ενώ τα κράτη-μέλη που είναι μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας, για αυτά η ΟΛΑΦ θα ερευνά συμπληρωματικά και σημερα ενω τα κρατη μελη που ειναι μελη της ευρωπαικης Εισαγγελίας, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν στενή και συνεχή συντονισμό ε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουμε θεσπίσει και ιδρύσει το Γραφείο Συνδέσμου στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο φυσικά είναι έδρα και του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Δικαστηρίου και πολλών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε το να έχουμε αποσπασμένους υπαλλήλου τη ΟΛΑΦ και στο Λουξεμβούργο θα βοηθήσει την καλύτερη συνεργασία όχι μόνο με τα θεσμικά όργανα στο Λουξεμβούργο, αλλά θα βοηθήσει τη συνεργασία και με τι ε, εθνικέ αρχέ του Λουξεμβούργου. Τέλο, λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι η υπηρεσία μα θα πρέπει να προσαρμόσει το ερευνητικό του έργο και στι νέε προκλήσει που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την στρατηγική από τον αγρό στο πιάτο και άλλου τομεί που λαμβάνουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οι μονάδε που προηγουμένω ασχολούνταν με απάτη στο εισόδημα και τις παραποίησεις έχουν ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό. Και μάλιστα σημαντικά περιστατικά όπως είχαμε με το λιγμένο γάλα σε σκόνη, το αλογίσιο κρέας και άλλα σοβαρά περιστατικά που αφορούσαν σκάνδαλα σε τρόφιμα ε, οδήγησαν σε επανειλημμένες εκκλήσεις για ενίσχυση του αντίστοιχου ερευνητικού μας έργου και την αντιμετώπιση ε, της πολιτικής ώστε να προστατεύει πραγματικά την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Με όλα αυτά κατά νου έχουμε τώρα μια ειδική μονάδα για τις έρευνες στο παράνομο εμπόριο, την υγεία και το περιβάλλον. Η Όλαφ ήταν ήδη ενεργή ε, στην καταπολέμηση επιστημιστικής απάτης και με επιτυχία έχει διερευνήσει τέτοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Η νέα μονάδα θα συνεχίσει να ερευνά τέτοιες υποθέσεις αλλά με πιο κεντρικό τρόπο Βάσει της εμπειρίας που είχαμε κατά την έρευνα περίπλοκων διασυνοριακών υποθέσεων και χρησιμοποιώντας τις ανα... αναλυτικές και εγκληματολογικές μας δεξιότητες που έχουμε αναπτύξει σε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας. Έχουμε ήδη διαπτά αποτελέσματα κατά την αντιμετώπιση απροσδόκητων προκλήσεων, όπως αυτό που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, για να προστατεύσουμε την την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε κίνδυνο από απατεώνες ε, που διέθεταν ακατάλληλες μάσκες ή ακατάλληλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Μάλιστα με τη νέα δομή θα μπορέσουμε πολύ πιο ενεργά να προστατεύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνεται καλύτερη ανάκτηση των αχρηστήτων καταβληθέντων. Επίσης, έχουμε αυξήσει τη, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πέραν αυτών που ίσχυαν για τους νέους ερχόμενους. Και μάλιστα το μαθησιακό πακέτο που έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόσει την αναδιοργάνωση της ΟΛΑΦ περιλαμβάνει ειδικέ ε, εκπαιδευτικές διαδικασίες για τις ερευνητικέ δραστηριότητες, για την αντιμετώπιση επιλογών και ειδικές, ε, ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μάνατζερ και καθοδήγηση για την αλλαγή και την μετάβαση. Εν κατακλείδη, με τη νέα δομή η ΟΛΑΦ θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για να προστατεύσει τον κοινοτικό προϋπολογισμό ακόμη πιο αποτελεσματικά και μέσω των ερευνητικών της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων για την πρόληψη της απάτης. Με τη νέα οργάνωση έχουμε ενισχύσει τη θέση μας και μπορούμε πλέον να αυξήσουμε τη συνεργασία με τους ε, πρωταρχικούς μας εταίρους και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να ξεχνούμε όμως και την Ευρωπόλ, την Eurojust και τις Εθνικές Αρχές. Πιστεύουμε ότι το ίδιο θα κάνουν και οι εταίροι μας και θα ε, ενισχύσουν τη συνεργασία τους μαζί μας. Αξιοποιώντας το έπακρο το δυναμικό της οργανωσής μας, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των πόρων μας. Όπως ξέρετε, η ΟΛΑΒ θα χάσει 45 θέσεις εν ώψη της ίδρυσης ε, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ενώ ο φόρτος εργασίας μας δεν πρόκειται να μειωθεί στο μέλλον. Οπότε θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και ιδιαίτερα την πρόεδρό της, την κυρία Χόλμαϊρ, που μας παρέχουν την αμέριστη υποστήριξή τους για το θέμα των πόρων ε, και για την έκκληση που απευθύνατε στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ζητήσατε επαρκείς πόρους για την ΟΛΑΦΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Εβίλε. Κύριε Γενική Διευθυντά, Έχουμε τον Γιάν Μούλτερ, ο οποίος έχει συνδεθεί μαζί μας, είναι ε, πρόεδρος της ε, Εποπτικής Επιτροπής. Γιάν, μας ακούς? Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε στην Επιτροπή μας λόγο σήμερα. Μας ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής για τις προθέσεις του και να πω ότι εμείς ως Εποπτική Επιτροπή συνεδριάζουμε μία φορά το μήνα και σε κάθε συνεδρίαση ενημερωνόμαστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στην υπηρεσία. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τις προθέσεις του Γενικού Διευθυντή. Δεδομένων των συνθήκων με τις νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αλλαγές του τομείς πολιτικής ήταν λογικό να υπάρξει αναδιάρθρωση. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να συνεργαστεί με το Γενικό Διευθυντή στενά και γι' αυτό θα πρέπει η συνεργασία να είναι καλή. Όπως και συμβαίνει για τον λόγο αυτό δεν υπήρξε κάποια διαφωνία ή κάποια αντίρρηση ε, ως προς την έγκριση της ε, αναδιάρθρωσης. Βέβαια το μέλλον θα δείξει τι θα γίνει, όμως σε αυτό το στάδιο εμείς ε, δεν έχουμε αμφιβολίες, ούτε είμαστε καχύποπτοι. Αυτά λοιπόν από την ε, Εποπτική Επιτροπή της Όλαφ. Are you still there? Είστε εκεί? Με ακούτε? Λίγο Μάριαν, του το Ο λόγος στο Μάριαν Μαρινέσκου. Δεν πρόλαβα να του δώσω το λόγο και έφυγε. Μάριαν, είσαι εδώ. Ελπίζω να μην φταίω εγώ που έφυγε. Αν βγάλεις το χέρι σου από το κουμπί μπορώ να μιλήσω. Διαφορετικά δεν μπορώ να μιλήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τον λόγο. Κύριε Ήταλα. Ελπίζω η αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σας να βοηθήσει το έργο σας, να σας κάνει πιο αποτελεσματικούς. Ο κανονισμός αυτός που βρίσκεται να εξελίξει και αφορά την συνεργασία Όλαφ και Ευρωπαϊκής Συγγελίας θα σας βοηθήσει να γίνετε πιο αποτελεσματικοί. Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ καλές και ελπίζω να καταφέρετε να περάσετε τις προτάσεις αυτές και όχι μόνο τις προτάσεις που αφορούν τα κράτη-μέλη, αλλά και εκείνες που αφορούν την ίδια την Όλαφ. Ακόμα και αν αυτές οι προτάσεις δεν χαροποιούν τους πάντες. Ελπίζω λοιπόν να στηρίξετε τη δουλειά που έχει γίνει πάνω σε αυτόν τον κανονισμό. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε συμφωνήσαμε εμείς, αλλά το Συμβούλιο δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες του. Και πιστεύω επίσης ότι η αναδιάρθρωση αυτή θα είναι προς όφελος της Όλαφ και των μελλοντικών της δραστηριοτήτων. η δραστηριότητα της υπηρεσίας θα πρέπει να αξιολογηθεί. να γίνει τόσο αξιολόγηση όσο και πρόληψη έτσι ώστε να εργαστείτε καλύτερα διότι είναι προτιμότερο να προλάβεις μια κατάχρηση παρά να κυνηγά αυτόν που έχει καταχραστεί. Έτσι υπερασπιζόμαστε καλύτερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Τώρα, για τα υπόλοιπα έχω να πω ότι ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα και να ολοκληρώσουμε το έργο μας για τη συνεργασία Όλαφ και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ελπίζω η συνεργασία αυτή να βελτιώσει πάρα πολύ ε, την αποτελεσματικότητά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάριαν. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου θερμά για ε, την, εσένα για την εξαιρετική δουλειά σου πάνω στον κανονισμό Όλαφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους ε, σκιώδης Τώρα έχουμε την Κατερίνα Κινίτσι στη γραμμή και έπειτα την Μισελ Ριβαζή, η οποία ήταν ιδιαίτερα δραστήρια ως σκιώδης και εργάστηκε σκληρά. Ελπίζω λοιπόν το Συμβούλιο να κάνει και αυτό τη δουλειά του και να ολοκληρώσουμε τις διαβουλεύσεις σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για την καλή συνεργασία και θα δώσω τώρα τον λόγο στην Κατερίνα Κινίτσι, η οποία νομίζω είναι μαζί μας από τη Σικελία. Καταρίνα. Sí, presidente. Mi... Super. Perfect. We can hear you. Perfect. Perfect. Grazie, Presidente. Intanto è davvero un piacere. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω και βεβαίως χαιρετίζω όλους τους παρόντες ε, στην αίθουσα αλλά και αυτούς που μας παρακολουθούν από τις οθόνες τους. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά το συντομότερο δυνατόν στο χώρο εργασίας μας. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τον Επιτρόπο Χάν αλλά και τους λοιπούς ε, ομιλητές. Όπως είπες αγαπητή Μόνικα και εγώ είμαι πεπισμένη ότι να αντιμετωπίσουμε την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά και για να εντοπίσουμε τη διαφθορά, είναι απαραίτητο να επικαιροποιούμε συνεχώς τα μέσα μας, τους πόρους μας, σε, και σε επίπεδο Όλαφ και σε επίπεδο των άλλων ε, οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών. Ο κανονισμός του Όλαφ είναι πολύ σημαντικό. Ε, τον έχουμε βελτιώσει του τελευταίου μήνε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους οι εισηγητές ε, που εργάστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, ενίσχυση λοιπόν των αρμοδιοτήτων της Όλαφ και εξασφάλιση ενός ορθού συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τους ε, κινδύνους που προκύπτουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλήσουμε και για την κατάρτιση αλλά και για τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη και με τις χώρες και ε, ε, το συντονισμό μεταξύ των χωρών που θα αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και αυτών που δεν θα συμμετέχουν στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες ακόμα, διότι είμαι πεπισμένη ότι το έργο της Όλαφ ε, εδώ μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σημασίας. Θα δημιουργήσουμε κάποια κέντρα γνώσεων, κέντρα αριστείας ε, για την καταπολέμηση της απάτης και γνωρίζουμε ότι στο προσεχές μέλλον, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στη διάθεση των κρατών μελών ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης φιλόδοξο για να βγούμε από την κρίση που έχει πλήξει όλες τις χώρες μας μετά την πανδημία της COVID. Ε, στη χώρα μου η εισαγγελία που αντιμετωπίζει τη μαφία ε, έχει, ε, ε, έχει αναφέρει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις να παρέμβουν και να επηρεάσουν το πού θα διατεθούν τα χρήματα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ε, ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ο κίνδυνος, ο ε, κίνδυνος παρίσφρησης αυτών των οργανισμών στη διαδικασία κατανομής των κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ε, το Νοέμβριο θα το έχουμε αυτό και βεβαίως θα χρειαστούμε την υποστήριξη της Όλαφ στην πρώτη φάση αυτή της έρευνας και θα πρέπει να υπάρχει ένας συνεχής συντονισμός καλό είναι ότι θα έχουμε μια νέα μονάδα με έδρα το Λουξεμβούργο, έτσι ώστε να έχουμε στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι επίσης απαραίτητο να ξεκινήσει αυτή η συμφωνία συνεργασία μεταξύ της Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι κρίσιμης κρίσιμη σημασία για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίε. Και δεν ξέρω εάν στα πλαίσια αυτή τη αναδιοργάνωση που είναι σημαντική, έχουμε ήδη σκεφτεί ε, ένα συντονισμό με την κυρία Κοβέζη, την καινούρια εισαγγελέα, έτσι ώστε να ε, εντοπίσουμε ποιοι είναι οι τομεί εκείνοι που υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο ε, ε, διαφθοράς, αλλά και, και μεγαλύτερος κίνδυνος ε, ε, εγκληματικών οργανώσεων. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι συμβαίνει με το συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών των εθνικών ε, και πώς θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες ε, για να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη διαφθορά και την απάτη. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους προσκεκλημένους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο που μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ε, αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της αναδιοργάνωσης της Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κάτριν θα μιλήσει στη θέση της Μαρτίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και τον κύριο Ήταλα που μας παρουσίασε τη νέα δομή της Όλαφ. Και εγώ έχω τις ανησυχίες που ανέφερε η κυρία Χολμάιερ ε, σε αυτήν την κρίσιμη εποχή, την δύσκολη οικονομική εποχή ε, βλέπω ότι θα υπάρξει περικοπή του προπολογισμού ε, της Όλαφ. Αν είχε μείνει μαζί μας ο κύριος Χάν θα τον είχα, θα τον είχα προτρέψει τις επόμενες εβδομάδες διαπραγμάτευσης τουλάχιστον ε, να κάνει μια προσπάθεια να ε, διαφυλάξει τη δυνατότητα που έχουμε ως Ευρώπη να ελέγχουμε τα δημοσιοοικονομικά μας. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν διαθέτει τεράστια ποσά ε, με πιο απλές προϋποθέσεις ε, για την ανάκαμψη και πολύ καλά κάνει. Όμως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε εκεί που πρέπει. Γι' αυτό και ο ρόλος της Όλαφ ε, είναι κρίσιμος. Ε, έχω κάποια ερωτήματα προς τον κύριο Ήταλα. Εσείς θεωρείτε ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των δυνατοτήτων ε, τη Όλαφ για να μπορέσει να επικεντρωθεί στι χώρες εκείνες που δεν αποτελούν μέρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, και όπου ενδεχομένως να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ε, δημοσιονομική, απάτης, οικονομικής απάτης. υπάρχει ένα ειδικό πεδίο που αφορά τις χώρες αυτές, ένα ειδικό πεδίο έρευνας για τις χώρες αυτές. Επίσης, πώς θα επηρεαστεί η επιλογή των υποθέσεων προς τη διερεύνηση, θα αλλάξει αυτό Επίσης πιστεύετε ότι οι έρευνες θα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Ε, πώς, ποιος είναι ο αντίκτυπος. Για μια φορά πάντως θέλω να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε αυτό το εξαιρετικό έργο. Η Επιτροπή σας ε, η Επιτροπή μας θα είναι πάντα αρρωγός στις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Μίσελ Ριβαζή έχει συνδεθεί μαζί μας και ελπίζω να μπορέσουμε να την ακούσουμε. suis la Ναι, πολύ ωραία. Ε, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ κυρία Ήταλα για την παρουσίαση. Εγώ είχα κάποια ερωτήματα, διότι βεβαίως υποστηρίζω με φανατισμό την Όλαφ ε, και θέλω να υποστηρίζω και τον συνάδελφο τον κύριο Μαρινέσκου για το έργο του, που ήταν σημαντικό πολύ σημαντικό, δεν αναφερθήκατε στην παρουσίασή σας του οργανιγράμματος για τον ρόλο του ελεγκτή. Ξέρετε ότι οι βουλευτές ζήτησαν να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεγκτής. Ε, έμαθα ότι αυτός ο ελεγκτής τελικά θα εξαρτάται διοικητικά, θα συνδέεται διοικητικά με την Επιτροπή Παρακολούθησης της Όλαφ, εμείς θέλαμε να είναι απολύτως ανεξάρτητος από την Όλαφ, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, από την Κομισιόν. Τι συμβαίνει τελικά. Ε, δεύτερο ερώτημα. Έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητές σας σε ό,τι αφορά την απάτη, ε, τη διατροφική, που είναι τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα μετά τη στρατηγική αυτή από το αγρόκτημα ε, στο πιάτο, ε, για πόσους ανθρώπους μιλάμε τελικά, περισσότερους δηλαδή ανθρώπους προσωπικό που θα ασχοληθεί με αυτή τη μορφή απάτης. Κάτι άλλο, δεν υπάρχει πια ένας μηχανισμός ε, επεξεργασίας των προσφυγών και αυτό μου προκαλεί έκπληξη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσες, πόσα, πόσους φακέλους εξετάσατε, ποια είναι η φύση των φακέλων αυτών. Στην έκθεση λοιπόν δραστηριοτήτων σας, την ετήσια, ε, και αυτό το ερώτημα πάει και στον κύριο Μίλλερ ε, στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Μπορεί να έχουμε ένα κατάλογο των προσφυγών. Είναι σημαντικό για μας τους ευρωβουλευτές να γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι ο αριθμός των προσφυγών που έφτασαν στην Όλαφ, την φύση των προσφυγών αυτών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του ζητήματος της διαφθοράς. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση λοιπόν στα δεδομένα αυτά, όχι στι τελικέ εκθέσει για όλε αυτέ τι προσφυγέ, αλλά για την φύση τουλάχιστον των προσφυγών, που, ε, τον τόπο του και την, τον τύπο ε, διαφθορά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί ο ρόλο τη Όλαφ εδώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέτρης Σάβαρμα έχει το λόγο. Α, όχι και ο κύριος Κούς. Κύριε Κούς, πολύ σύντομα, γιατί μετά έχουμε το θέμα με την ΕΤΕΠ και δεν μπορούμε να δώσουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ήταλα για την παρουσίαση. Θα ήθελα με την ευκαιρία να θυμίσω ε, βεβαίως εδώ δεν υπάρχουν μέλη ε, που ήταν εδώ ε, πριν από τον κύριο Ήταλα, όταν ήταν εδώ μάλλον ο, ο, ο προκάτοχος του κύριου Ήταλα. Η μόνη καλή θυμάμαι. Ε, βέβαια, σωστά, ήταν και εσείς μέλος είσαστε. Ναι, θα θυμάστε λοιπόν τι συνέβαινε προκατόχου του κυρίου Ήταλα. Ήθελα λοιπόν να πω, να το πω έτσι και επισήμως, ότι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ήταλα και εδώ θα είμαι πολύ προσεκτικό στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω, έτσι, διότι έφερε την Όλαφ πίσω σε μια κάποια κανονικότητα. Και, όσοι θυμούνται καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ευχαριστώ γι' αυτό και το ερώτημά μου είναι το εξή: Με τη νέα οργάνωση, την αναδιάρθρωσή σας, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικές δυσκολίες, οι πιο μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε. Ίσως να μην έχει σχέση αυτό με τη νέα οργάνωση, αλλά μπορεί και να έχει. Ε, καλό θα είναι να γνωρίζουμε εμείς, τα μέλη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, ε, πώς βλέπετε εσείς το προσεχές μέλλον, στο προσεχές μέλλον ε, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι ε, οι δυσκολίες, οι κεντρικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε. Μάλιστα. Ο κύριο Κούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κούς. Ε, σα ευχαριστώ. Συνεχίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα, κύριε Ήταλα. Όταν ξεκίνησε ένα διάρθρωση δεν γνωρίζατε ε, εάν θα υπάρχει ταμείο ανάκαψή, τι θα γίνει, εάν αυτό το ταμείο θα ανέρχεται στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Ε, θεωρείτε πως ε, θα υπάρχουν και 70% περισσότερες περιπτώσεις απάτης. Τι θα κάνετε, θα τα βγάλετε πέρα με το προσωπικό που έχετε. Μα ανησυχεί πολύ. Εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας ε, διευκολύνουμε στο έργο σας, διότι αυτή η αύξηση προϋπολογισμού φαντάζομαι και φοβάμαι ότι θα σημαίνει και αύξηση δουλειάς για εσάς. Ευχαριστώ. Ωραία, θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στο όνομα της Επιτροπής Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ απολύτως ε, με την ανάλυση των Ευρωβουλευτών ότι υπήρξε μια ε, ριζική αλλαγή στην προσέγγιση της Όλαφ. Η Όλαφ έχει μια παράδοση να μην ακούει το προσωπικό και όπως δείχνει και η σχετική μελέτη είχαμε ανησυχητικά αποτελέσματα στη μελέτη αυτή, διότι η Όλαφ, το προσωπικό του Όλαφ ε, δεν ενθαρρυνόταν παρκώ ε, για να κάνει τη δουλειά του, δεν ε, εμπλεκόταν αρκετά στο, στις αποφάσεις. Γενικά, η Γενική Διεύθυνση δεν είχε μια κουλτούρα καινοτομία και αλλαγών και αυτό ήταν κρίμα διότι οι συνάδελφοι είχαν εξαιρετικέ δεξιότητε. Χαιρόμαστε λοιπόν που υπάρχει τώρα μια πιο συμμετοχική προσέγγιση, η οποία είναι παραδειγματική για όλε τι μελλοντικέ οργανώσει. Καλούμε του συναδέλφου τη Γενική Διεύθυνση ε, μάλιστα ανθρωπίνων πόρων να λάβουν γνώση για όλε τι μελλοντικέ αναδιοργανώσει. Συχνά το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει αναδιοργανώσει που έχουν επιβληθεί χωρί κάποια διαβούλευση με του συναδέλφου, χωρί ε, ε, συζητήσεις, ενώ στην περίπτωση της Όλαφ είχαμε για εβδομάδες συναντήσεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε μια συνδιαχείριση, έτσι. Θέλουμε απλώς ε, να εκμεταλλευτούμε τη συνεισφορά των συναδέλφων. Επίσης είναι δύσκολο για την ώρα να ε, αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα αυτής, αυτού του εγχειρήματο. Ως Επιτροπή Προσωπικού πάντως εμείς σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια έρευνα ε, ικανοποίηση των συναδέλφων για να μας πούν πώς το βλέπουν και βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα, θα σας διαβιβαστούν. Τα δύο μόνο ανησυχίες που υπάρχουν είναι η έλλειψη σαφήνειας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Όλαφ και Εισαγγελίας. Οι συνάδελφοι της Όλαφ έχουν την εντύπωση ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί. Το έλαβα και στα συμπεράσματα του σεμιναρίου που έλαβε χώρα κάποια στιγμή. Υπήρχε ο, χρο, κίνδυνος ο Όλαφ να περιθωριοποιηθεί. Αυτή η ανησυχία ότι θα περιθωριοποιηθεί ο Όλαφ λόγω της αγγελίας. Η δημιουργία αυτού του μικρού γραφείου τριών ατόμων στο Λουξεμβούργο είναι χρήσιμο βήμα. Κάποιοι βεβαίως αν αναρωτιούνται κατά πόσο είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Θα χρειαστεί να υπάρχει μια βούληση συνεργασίας ε, την οποία εμεί υποστηρίζουμε. Το δεύτερο η δεύτερη ανησυχία είναι οι πόροι. Ε, ανησυχούν οι συνάδελφοι ότι οι πόροι δεν θα είναι στο ύψο ε, των προκλήσεων. Αυξάνονται ε, οι ευθύνε, ε, αυξάνονται τα καθήκοντα, αλλά δεν αυξάνονται οι πόροι. Αυτό ε, συμβαίνει γενικότερα στην Κομισιόν βέβαια, αλλά ειδικότερα και στην περίπτωση της Όλαφ. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής αυτής για τη δουλειά που κάνει σε ένα ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα την κατεπολέμηση του, ε, της παρενόχλησης. Ήμουν και στη συνάντηση ε, στην ΕΟΚΕ. Είναι προφανέ ότι μόνο χάρη σε εσά και στην ε, Όλαφ μπόρεσαν να απαντηθούν σχετικέ ε, διαματρίες και προσφυγέ. Θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μα γι' αυτό. Εσεί η Όλαφ και ο Όμπουτσμαν, ο διαμεσολαβητή, είναι οι πραγματικοί ε, παράγοντες κλειδιά για να θέλουμε να έχουμε μια πολιτική μηδενική ανοχή απέναντι στην παρενόχληση. Διότι πολύ συχνά έχουμε μια πολιτική μηδενική πολιτική βούληση για την καταπολέμηση ε, της παρενόχλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς για το έργο σας και τη δουλειά που έχετε κάνει. Ως απάντηση στα πολύ καλά σας λόγια, να πω και εγώ ότι και εμείς είμαστε πεπισμένοι για το αποτελεσματικό σας έργο και θέλουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ε, είναι εξοργιστικό κάπως ε, το να παρατηρούμε ότι κάποια κράτη-μέλη συνεχίζουν να δημιουργούν εμπόδια και τα κράτη αυτά μάλιστα είναι εκείνα που έχουν τους περισσότερους λόγους να στηρίζουν την Όλαφ και το έργο της. Είναι εκνευριστικό αυτό, όμως ε, θα συνεχίσουμε τη δουλειά και δεν θα μας πτωίσει. Αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στον Ματίας Βίλ Όχι, στον κύριο Ήταλα. Στον κύριο Ήταλα για τα καταληκτικά του σχόλια. Για ενδεχόμενες ερωτήσεις, ε, κύριε Βίλ, ε, είστε διαθέσιμος. Δεν είχε βέβαια κάποιος ευρωβουλευτής ε, κάποια ερώτηση να θέσει, όμως είναι καλό που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ήταλα, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους Ευρωβουλευτές για τις πολύ εύστοχες και συμπαντικές ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να καλύψω όσες περισσότερες γίνεται. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανάκαμψης, τεράστια πρόκληση για όλους μας. Για όλους μας και για την όλα φυσικά. Αυτό δεν το γνωρίζαμε όταν ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση. Δεν γνωρίζαμε την έλευση του σχεδίου ανάκαμψη. Αλλά νομίζω ότι με την νέα διοργάνωση είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέε προκλήσεις. Γιατί τώρα είμαστε πολύ πιο ελαστικοί και ευέλικτοι. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό στο πακέτο ανάκαμψης είναι ότι ε, φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπιστεύεται και τα ελεκτικά συστήματα στα επιμέρους κράτη-μέλη. Αλλά θέλουμε και ένα πιο κεντρικό σύστημα, να μπορεί και η Όλαφ να ασκεί κάποιες έρευνε. Θα σταθώ στα πιο σημαντικά σημεία. Υπάρχουν πολλά, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα ε, και να χορηγούν τις πληροφορίες ε, που ζητάμε για τους δικαιούχους των κονδύλιων για τους τελικούς χρήστες και δικαιούχους. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε τους τελικούς χρήστες, πώς θα κάνουμε την έρευνά μας. Και σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων, δεν είναι δυνατόν να φανεί ο τελικός χρήστης. Οπότε είναι σημαντικό, από τη στιγμή που τα χρήματα θα πάνε στα κράτη-μέλη, να συγκεντρώνουν αυτές τις πληροφορίες και να τις δίνουν στις ερευνητικές αρχές. Επίσης, τέθηκε η ερώτηση για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την ΕΠΟ. Με τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις έχουμε καθημερινή επαφή και γίνεται σε πολύ καλό κλίμα αυτή η συνεργασία γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε πολλά κοινά και κοινέ δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε. Το σημαντικό εδώ είναι ανοιχτή και διαφανής ανταλλαγή ε, πληροφοριών και με τη Europol και με τη Eurojust, γιατί όλοι δραστηριοποιούμαστε στον ίδιο τομέα και αν δεν ανταλλάσσουμε πληροφορίες, τότε δεν θα είμαστε ε, αποτελεσματικοί ούτε ημένου ούτε είδε. Και ό,τι οργάνωση και αν έχουμε, δεν θα μας καλύψει αν δεν είμαστε όλοι ανοιχτοί και διαφανείς στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής, έχουμε μια ειδική μονάδα που κάνει τις επιλογές και τις κάνει και πολύ καλά. Και φυσικά έχουμε και κοινέ προκλήσεις για το πώς θα το κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά είμαστε καλά προετοιμασμένοι γιατί όλοι είμαστε επαγγελματίε και είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε καλά. Τώρα, έχουμε και την έθεση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για να γίνονται γκέρος οι έρευνες Φυσικά υπάρχει πάντα το θέμα των πόρων. Ε, χάσαμε 45 θέσεις στην ΟΛΑΒ. Μπορεί να έχουμε έναν ε, ε, ερευνητή που μιλά μια γλώσσα που χρειάζεται, αλλά αν είναι ένας μόνο αρμόδιος και είναι σε αναρωτική, τότε δεν έχουμε κανέναν που θα μιλά τη γλώσσα που χρειαζόμαστε. Τι θα πάμε στο Google Translate για να κάνουμε τις ερευνές μας. Αν αρρωστήσει ο αρμόδιος ε, ανακριτής ε, και έχουμε μόνο έναν. Επίσης, υπάρχει και το θέμα του ελεγκτή. Ο ελεγκτής ε, που θα προσθεθεί στη γραμματεία. Και στον τριμερή διάλογο θα δούμε το αποτέλεσμα του συμβιβασμού και πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Τώρα, για τις καταγγελίες. Πέρσι είχαμε 8, αν δεν κάνω λάθος, και πρόπερσι 7 καταγγελίες, οπότε δεν έχουμε τόσες πολλές καταγγελίες. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με, τον, ε, με το διορισμό του ελεκτή. Ήταν πρώτα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οριστεί ένας ελεκτής. Αλλά ούτως ή άλλως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι από τις πιο από τα θεσμικά όργανα στον κόσμο που υφίστανται τους περισσότερους ελέγχους. Έχουμε το ελεκτικό συνέδριο, έχουμε τους εσωτερικούς ελεγκτές, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου, τον Διαμεσολαβητή, το Δικαστήριο, την Εποπτική Επιτροπή που συνεδριάζει κάθε μήνα. Και τώρα θα προσθεθεί και ένας επιπλέον ελεγκτής. Οπότε από ελέγχους άλλο τίποτα. Νομίζω ότι έχουμε τους περισσότερους ελέγχους. Αλλά είναι λογικό να υπάρχουν τέτοια έλεγχη σε ένα όργανο που έχει τέτοιες ε, ερευνητικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ο κύριος Σαρβαμά ρώτησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πώς τις βλέπουμε. Μία πρόκληση είναι η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη Europol και τη Eurojust. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές τις υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό. Και επίσης, ε, πόσο, τι κίνητρα θα δώσουμε στο προσωπικό. 45 θέσεις τις δώσαμε από την ΟΛΑΒ στην ΕΠΟ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ακούστηκαν κάποιες φήμες ότι θα πρέπει να δώσουμε και άλλες θέσεις. Μα πώς ε, θα κινητοποιήσουμε το προσωπικό μας να κρατήσει τον ενθουσιασμό του και την προσήλωσή του, γιατί ήδη υπάλληλοι μας δεν έχουν Σαββατοκύριακα, νυχθημερών οργάζονται και τώρα θέλετε να παραμείνουν ε, ενεργοί και ενθουσιασμένοι όταν απειλούνται και με περαιτέρω μείωση προσωπικού. Πάντως χαίρομαι που ομόφωνα η Επιτροπή σας Μα υποστήριξε και υποστήριξε το προσωπικό και του υπαλλήλου. Μα Είναι πολύ σημαντικό για το δικό τους ηθικό. Τώρα, είμαστε μόνο 83. Μεγάλη πρόκληση. Εκτιμώ το έργο του εισηγητού και εσεί, κυρία Πρόεδρε ήσταν παρούσα. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε καλή συμβαστική λύση δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα πάντα, αλλά ούτε για το Κοινοβούλιο ούτε για το Συμβούλιο. Αλλά αυτό το νόημα έχει ο συμβιβασμό. Κανεί δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο. Τώρα, αν το Συμβούλιο θέλει να ξανανοίξει αυτό το θέμα με την πρόσβαση στου τραπεζικού λογαριασμού και αν ε, λάβετε και εσείς απόφαση για το τι θέλει το Συμβούλιο, να μπει σε μια αιτιολογική σκέψη αυτή η αλλαγή ότι η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα επιτρέπεται μόνο από εθνική διοικητική αρχή. Σε μερικές χώρες όμως δεν υπάρχει καν τέτοια αρμόδια διοικητική αρχή. Εμείς έχουμε μια εκρεμή υπόθεση σε μια χώρα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω πληροφορίες, αλλά η χώρα δεν μας δίνει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και κάποιες συμμορίες ήδη ενεργοποιούνται σε αυτή τη χώρα. Οπότε αν δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι σαν να δημιουργούμε φορολογικό παράδεισο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εγκληματίες και πρόσφορο έδαφος για τις συμμορίες για να ενεργοποιούνται. Ελπίζω λοιπόν να επιμείνετε στον τριμερή διάλογο να παραμείνει αυτή η συμβαστική πρόταση για την πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Γιατί αυτό που προτείνει το Συμβούλιο δεν είναι καν η τρέχουσα κατάσταση, αλλά είναι μια παλινδρόμηση σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Και αυτή είναι σημαντική πρόκληση. Να διαφυλάξουμε στους, στους τριμερείς διαλόγους την συμβαστική λύση στην οποία έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Όλαφ έχει τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Όπως σας είπα, σεβόμαστε απόλυτα το έργο σας. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό Διευθυντή και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει και εκείνη την Όλαφ. Ελπίζω να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά με κράτη-μέλη. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στο έργο σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης και να ζητήσω να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ. Μετά από παράκληση της ΕΤΕΠ, θα πρέπει αυτό το κομμάτι να γίνει κυκλισμένο των θυρών. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση που δείχνετε. Και ζητώ συγγνώμη